Να αρχίσουμε. Προτείνω η κυρία Βαλενσιάνο δεν είναι εδώ για το πρώτο τμήμα και μου ζήτησε να προεδρεύσω εγώ. Εγκρίνουμε στο πρώτο σημείο το σχέδιο τη διάταξη. Ζητάει κάποιο τροποποίηση. Παντσέρι. Όχι. Αιδευτικό είναι το παντσέρι. Ε, θα πρέπει να εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά ε, της συνεδρίασης ε, που έλαβε χώρα στις 16 και 17 Ιουνίου. Ενστάσεις. Μπορούμε τότε να εγκρίνουμε το, το, τα πρακτικά και θα περάσω τώρα στις ανακοινώσεις μας. Το κοινοβούλιο μας, όπως το γνωρίζετε διότι πολύ ενδιαφέρονται για αυτό του είδους τις ε, δραστηριότητε. Ενέκρινε τρία ε, κατεπίγοντα ψηφίσματα στην Ολομέλεια της, ε, του Σεπτεμβρίου για τη Ρωσία, για τις περιπτώσεις Έστον Κόβερ, Όλεξ Αντσόφ και Αλεξάνδρ Κολτσένκο, ένα δεύτερο για την Αγγόλα και ένα τρίτο για το Ζαρμπαϊτζάν. Το τρίτο συζητήθηκε εκτενώς γιατί οι Αζέροι αποφάσισαν να αποσυρθούν από την ε, διακοινοβουλευτική γεωρονέστη. Μετά, δεύτερη ανακοίνωση για το βραβείο Ζαχάροβ 2015. Έχουμε διαφόρους υποψηφίους για το 2015. Στις 10 Σεπτεμβρίου την 5η ε, ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι παρουσιάσεις θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Δευτέρα, στην ε, κοινή συνεδρίαση Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης ε, και της δικής μας Υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αναφέρω τα ονόματα απλώς. Θα γίνει παρουσίαση τη Δευτέρα, 10 λεπτά ε, για τον καθένα. Ραΐφ Μπανταουί, ένας ε, blogger από το Σουδάν, έχει καταδικαστεί σε κάθε εξή δεκαετή και ε, χίλια... Ε, και χίλια μαστιγώματα ε, επειδή ε, για την ιστοσελίδα ε, Free Sound Liberals στη συνέχεια πολιτική κρατούν από τη Βενεζουέλα καθώς και δημοκρατική αντιπολίτευση της τράπεζας της Δημοκρατικής Ένωσης για την διατρόντιφρόντος λοιπόν εναντίον του Χούγκο Τσάβες, Έτνα Ντάν Ισμαήλ από τη Σομαλία, είναι πρώην υπουργό, αγωνίζεται για, κατά ε, τη, του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων ε, και έχει ε, ιδρύσει την κλινική Έτνα Άνταν στην Αργίσα στη Σομαλία. Μπόρις Νεμτσόφ, πρώην πρωθυπουργό και ο οποίος δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο στη Μόσχα. Νάντια Σαφτσέγκο είναι η πιλότος από την Ουκρανία, μέλος της ΡΑΝΤΑ και ε, του, ε, της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης συνελήφθη στις 18 Ιουνίου και μεταφέρθηκε παράνομα στη Ρωσία και είναι φυλακισμένη και παραμένει εκεί περαστή συνέχεια Edward Snowden ο Αντουάν Ντελτούρ από την PricewaterhouseCoopers και η Στεφανή Ζιμπό, ε, η οποία έκανε αποκαλύψεις για την εφοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος για την Ελβετική Τράπεζα UBS AG. Αυτή είναι η υποψήφοι και στην, Μικτή Επιτροπή, στην κοινή συνεδρία των τριών επιτροπών τη Δευτέρα θα παρουσιαστούν οι υποψηφιότητες. Θα ήθελα τώρα να σας πω και κάποια πράγματα για την αντιπροσωπεία Ντρουά που θα μεταβεί στη Σερβία στο Βελιγράδι πιο συγκεκριμένα από αύριο το πρωί μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Είναι μια κοινή αντιπροσωπεία, μεικτό κλιμάκιο δηλαδή με την ΑΦΕΤ. Σήμερα το βράδυ φεύγουμε για να γίνει μια αποτίμηση της κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή την χώρα υποψήφια για την προσχώρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατο προσφυγικό πρόβλημα η Σερβία για ε, τα μέλη της Επιτροπής μας, ε, Λάσλο Τέκες, Αντρέ Κόβατσεφ και Σωράη Αγώστα. θα είναι τα τρία μέλη της Επιτροπής μας ε, και άλλοι θα ε, μεταβούν εκεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα μεταβούν και εκείνοι στη Σερβία και μην ξεχνάμε θα πάνε και μια μέρα στο κοσφόπεδιο. Αυτά για τις ανακοινώσεις τώρα. Σημείο 4 είναι απολογισμός ε, πεπραγμένων από τις αποστολές μας στο Ισραήλ. Ο συνάδελφος Γιώσεφ Βάιντενχόλσερ ε, ηγήθηκε αυτής της αντιπροσωπείας ε, στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα στην Παλαιστίνη από τις 20 μέχρι 24 Ιουλίου στις αρχές των καλοκαιρινών διακοπών. Πέντε ημέρες κράτησε η επίσκεψη. Συναντηθήκατε με μέλη του νομοθετικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου και με μέλη της ΕΚΝΕΣΕΤ, με ειδικού εκπροσώπους της κυβέρνησης και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Δεν κατέστη δυνατόν να πάμε στη Γάζα, ε, όμως ε, επισκεφθήκανε πολλές ε, πόλεις και χωριά στο Ισραήλ και στην ε, Δυτική Όχθη για να ε, μελετήσουν ε, εντελεχώς την κατάσταση. Έχει μοιραστεί το σχέδιο έκθεσης της αποστολής. Είναι πληρέστατο, 27 σελίδες και παραρτήματα. Έχουμε τον κύριο Μπόσακ εδώ ε, με βιντεοδιάσκεψη. Είναι ο διευθυντής της ε, Ούρνερα στη Γάζα που μπορεί να μας δώσει τη... να μας κάνει την ενημέρωση για την κατάσταση. Σε τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα μας ακούτε. Νομίζω ότι μας ακούτε. Βεβαίως σας ακούω ξεκάθαρα κιόλας. Πολύ ωραία. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Γιώσεφ Βάιτενχόλσερ, τον πρόεδρο της, ε, του κλιμακίου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη. Κύριε Βάιτενχόλσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε κάναμε μια αρκετά εκτενή έκθεση την οποία έχουμε δώσει. Ε, θέλω να και τη Γραμματεία για την εκπόνηση αυτής της ε, έκθεσης. Είναι γνωστή η ουσία της ε, ε, επίσκεψής μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι μας. Έχουμε συγκεντρώσει πολλές εντυπώσεις, οι οποίες βέβαια επηρεάζονται και από το πολιτικό κλίμα. Αυτό ήταν και ο στόχος του ταξιδιού μας, να μπορέσουμε να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση εκεί. Μπορούμε να πούμε ότι από τη μία πλευρά από την πλευρά των Παλαιστινίων υπάρχει μια, ένα κλίμα απόγνωσης, έλλειψης ελπίδας από την πλευρά της, του Ισραήλ υπάρχει κάποια σύγχυση γιατί υπήρξαν πολλές νέες εξελίξεις με τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης με την συμφωνία με το Ιράν και γενικά με την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τις εκτιμήσεις των υπευθύνων στο Ισραήλ. Θεωρούν λοιπόν ότι δεν τους ε, υποστηρίζει ε, κανείς για να κάνουν τις συζητήσεις με τους ε, συνομιλητές τους και ζητούν από εμά ως κοινοβουλευτικούς να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε σε αυτό το εγχείρημα. Κάναμε πολλές επαφές και συζητήσεις με εκπροσώπους της κυβέρνησης, με ΜΚΟ, κάναμε μια σειρά από επισκέψεις. Εμείς μπορέσαμε να κάνουμε πολλές ερωτήσεις στα άτομα αυτά, να έχουμε μια κριτική ανταλλαγή απόψεων πήραμε από ορισμένου συγκεκριμένε απαντήσει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ θετικό και είναι μια βάση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε στο μέλλον τη συνεργασία μας. Συζητήθηκε και το θέμα της κατάσταση στη Γάζα για τις στρατιωτικές επίσης του Ισραήλ. Μας ε, ανέφεραν κάτω από ποιες συνθήκες ο Γενικό Εισαγγελέα του Ισραήλ πώ αντιμετωπίζει το Ισραήλ μαζί με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο θέματα τα οποία έχουν προκύψει από την επέμβαση στη Γάζα. Σε ανοιχτό κλίμα όλα αυτά. Από την πλευρά του Ισραήλ βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν εντάσεις με ορισμένους που συναντήσαμε από τη λίστα την αραβική που κατέβηκε στις τελευταίες εκλογές θέλανε να υπάρχει κάποιος υπάλληλο από την Κνεσέτ ο οποίος θα παρακολουθήσει αυτές τις ε, συζητήσεις. Εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο ήταν το πιο ουσιαστικό και το οποίο επεσκίασε τα υπόλοιπα θέματα είναι το θέμα των επικισμών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο όλων των προσπαθειών να επιληθεί το πρόβλημα Βέβαια συνεχίζεται η πολιτική αυτή του επικισμού και διαιωνίζεται κατά κάποιο τρόπο, οπότε τίθεται ένα αμφιβόλο το θέμα της κυριαρχίας ενός ενδεχόμενου Παλαιστινιακού κράτους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι σαν ελβετική γραβιέρα να ασκήσει κανείς κυριαρχία και επομένως όλη αυτή η πολιτική επικισμού του Ισραήλ ουσιαστικά είναι μια αντιπαράθεση με τους Παλαιστίνιους και οδηγεί σε κάθε είδους τρευλώσεις. Και φυσικά βλέπουμε ότι οι Ισραηλοί έχουν σχεδόν απεριόριστο δικαίωμα να επικίσουν όποιες περιοχές θεωρούν χρήσιμος και να οικειοποιηθούν πόρους και κυρίως είδωρ στις περιοχές αυτές, φυσικούς πόρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να παρακολουθήσουμε την κατάσταση αλλά συγχρόνως πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο Ισραήλ τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται να περιοριστεί η δυνατότητα δράσης των ε, ΜΚΟ. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ για το κατά πόσο μπορούν να παίρνουν υποστήριξη από το εξωτερικό ΜΚΟ Εμείς ε, έχουμε διάφορους φορείς οι οποίοι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Παλαιστινιακή πλευρά υπάρχουν προσπάθειες να περιοριστεί ο ρόλος των ε, ΜΚΟ. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας. Και μια τελευταία παρατήρηση. Για την ε, πολιτική κατάσταση. εγώ βλέπω, η εντύπωσή μου είναι ότι ο χρόνος για μια πολιτική λύση σιγά σιγά εξαντλείται. Ήρθα σε επαφή με τον κύριο διαπραγματευτή των Παλαιστινίων. Προσπαθώ να βλέπω τον πρόεδρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολλοί πια οι Παλαιστίνοι οι οποίοι δεν βλέπουν καμία δυνατότητα λύσης και κινούνται περισσότερο προς ριζοσπαστικές κινήσεις. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δώσουμε μια νέα όθηση στην επίλυση του προβλήματος. Τις ε, λεπτομέρειες βέβαια θα τις βρείτε στην έκθεσή μας και έχουμε και δώσει και μια ανακοίνωση μια σύντομη ανακοίνωση τύπου η οποία περιλαμβάνει τα κυριότερα στοιχεία, αλλά αν θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση και φυσικά σταματάω εδώ για να δώσω και στους συναδέλφους να προσθέσουν αν θέλουν κάτι σε αυτά που είπα. Σας ευχαριστήσουμε και η κυρία Κουίστρ Ντοροβόλη είναι εδώ πέρα και μπορώ να της δώσω το λόγο να συμπληρώσει κάποια πράγματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Χόλτζα σας έχει δώσει αρκετές πληροφορίες για την αποστολή μας στο Ισραήλ και αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι απλώς να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν διοργανώσει, διοργάνωσαν αυτή την επίσκεψη, τους συνεργάτες και τους συμβούλους μας εδώ. Δεν νομίζω ότι ήταν μια εύκολη αποστολή, αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να πω. Και εγώ Συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ και εγώ νομίζω ότι γύρισα χωρίς καμία ελπίδα. Μιλώντας με νέους πολιτικούς, τους ε, ηλικιωμένους ξέρουμε ότι είναι ήδη αγγυλωμένοι στις απόψεις τους, αλλά και οι νέοι πολιτικοί είχαν ήδη αρκετή δυσπιστία σε εμάς, έθεσα πολλές φορές το ερώτημα, με ποιο μπορείτε εσείς από την άλλη πλευρά να έχετε μία επαφή, να φτιάξετε κάποια συνεννόηση. Είπανε, ναι μπορούμε με τον α με το β, αλλά και μετά επανέλαβαν όλα αυτά, όλες αυτές τις προκαταλήψεις και τις ε, απόψεις που γνωρίζουμε. Επομένως, η γενική παρατήρηση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες στην τωρινή στιγμή Είχαμε πολλές ε, επιμέρους συζητήσεις, πολλές επιμέρους εμπειρίες, αλλά γενικά έχουμε πάρει μια καλή επισκόπηση της κατάστασης. Νομίζω ότι πήραμε πολύ καλές πληροφορίες από άλλες τις πλευρές και συζητήσαμε τόσα πολλά σημεία που βέβαια θα άξιζε τον κόπο σε μια ειδική επίσκεψη το καθένα από αυτά να τα εμβαθύνουμε. Και φυσικά συζητήσαμε για το τι είδου μήνυμα θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω, τι θέλουμε να πούμε στην ανακοίνωση τύπου που θα δώσουμε. Ανεξάρτητα από την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο καθένα από εμά, νομίζω ότι ένα κοινό στοιχείο που πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν ήμασταν μια εξεταστική, μια ερευνητική επιτροπή. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε αυτό τον ρόλο. Μείναμε σε επιφανειακό επίπεδο και επομένως είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη κρίση για την κατάσταση <clears throat> στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω. Γνωρίζετε τώρα ότι έχουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα των προσφύγων στην Ευρώπη. Έχουν φτάσει πια και στο κέντρο της Ευρώπης. Επιτέλους θα μπορούσα να πω έχουν φτάσει και στο κέντρο της Ευρώπης. Αν, είναι κανείς, αν βρεθεί κανείς στο Ισραήλ βλέπει όλη αυτή τη γεωπολιτική κατάσταση με ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Το γεγονός ότι όπως είπε ο κ. Βαντεν Χόλτσερ οι Παλαιστίνοι νιώθουν απελπισία, δεν έχουν καμιά ελπίδα. Από την άλλη πλευρά λένε οι Ισραηλοί ότι αυτή τη στιγμή απαιτείται, απειλείται συγγνώμη, η ασφάλειά τους και βρίσκουν ότι είναι σε μια περιοχή του κόσμου η οποία είναι επικίνδυνη για αυτούς, <clears throat> γι' αυτό για μας το συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να αποκομίσουμε και το οποίο είναι κάτι το οποίο βλέπουμε από όλη αυτή την <clears throat> διαδικασία ότι είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τα προβλήματα των προσφύγων γιατί αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει σε μια λύση εκεί. Η ημέρα μας ήταν πολύ γεμάτη, πολλές φορές ξεκινούσαμε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ήταν πολύ κουραστικό, αλλά εντάξει ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, κάναμε πολλά πράγματα σε λίγες μέρες και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να έχουμε περισσότερες επαφές και πληροφορίες για τα θέματα αυτά. Αλλά υπήρξε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στην αντιπροσωπεία, συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα και είχαμε ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα διότι θέλουν και άλλοι βουλευτές το λόγο. Η κυρία Άουκεν. Ναι, με συγχωρείτε, μια σύντομη ερώτηση. Γιατί μόλις τώρα είδα τη δημοσίευση. Με εξέπληξε τον Ιούλιο, μετά την επίσκεψη. Ήμασταν εκεί με αντιπροσωπεία από τους Πρασίνους, περίπου ταυτόχρονα με σας. Αλλά αυτό που με ευνηδίασε είναι ότι η κατοχή αναφέρθηκε με μία μόνο μνήα έκκληση για άρση της ε, κατοχής αυτό γιατί δεν την παρατηρήσατε ή έχετε την αίσθηση ότι πρόκειται ε, για ισότιμη συνεργασία μεταξύ κατεχομένων και κατεχόντων. Πραγματικά με εξέπληξε που η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν ε, μίλησε για την κατοχή και την αναστολή της. Προέδρε Ρόβολ, δεν είμαστε οι πράσινοι και εξήγησα ότι είχαμε επανειλημμένως διαπραγματεύσεις με όλες τις πλευρές όμως δεν εμβαθύναμε σε κανένα θέμα ε, τόσο πολύ αφού είσαστε εκεί ως πράσινοι, είχατε τη δική σας δημοσίευση στον τύπο, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε τη δική σας γραμμή. Ο κ. Ich habe das auch zu Beginn gesagt το είπα και στην αρχή ότι ήμασταν μια αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αποστολή όχι να υποκαταστήσουμε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ο στόχος μας είναι να ήταν να επισκεφτούμε και να συζητήσουμε με τους συνομιλητές μας για θέματα τα οποία είναι κεντρική σημασία στις πολιτικές, να μάθουμε τις πολιτικές εκτιμήσεις τους μέσα στο πλαίσιο αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό που λέει η κυρία Άουκεν περιλαμβανόταν στην αποστολή μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέρκερ έχει ζητήσει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Βάιντεν Χόλτσερ και την κυρία Κούστο Τροβόλ. Είναι πραγματικά η σύγχυση στο Ισραήλ και η απόγνωση από την πλευρά των Παλαιστινίων. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, αν μιλάμε για δύναμη κατοχής και κατεχόμενα εδάφη, θα πρέπει να μην ξεχνάμε τι ακριβώς έγινε με την ε, Λωρίδα της Γάζας. Έχουν εκδιώξει όλους τους ε, ε, Εβραίους από την Λωρίδα της Γάζας. Έχει καταληφθεί τελείως από τους Παλαιστινίους. Δεν υπάρχει καμία λύση, καμία δυνατότητα λύσης όταν ακυρώνονται οι προϋποθέσεις για την λύση. Το 2001 υπήρξε επίθεση κατά των Ισραηλινών με δεκάδες νεκρούς από το, την Ισραηλινή πλευρά, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία ενός τείχους. Και αυτό δείχνει γιατί δεν έχουν σταματήσει αυτές οι αντιπαραθέσεις. Οι Ισραηλοί έχουν απειληθεί με το να τους σπρώξουν ως τη Μεσόγειο, να τους διώξουν. Γι' αυτό πρέπει να υπερασπιστούν και αυτοί τον εαυτό τους. Έχουν μπει 2,6 δισεκατομμύρια στη λωρίδα της Γάζας 140 εκατομμύρια μονάχα από τη Σαουδική Αραβία. Τι γίνανε αυτά τα χρήματα για μένα. Νομίζω είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίδονται από τα αραβικά κράτη. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ η κατάλληλη στιγμή να μιλάμε για ε, κατακτητές και αυτούς οι οποίοι κατέχουν τα εδάφη. Εγώ θέλω να συγχαρώ την αντιπροσωπεία για αυτά τα οποία ε, μας έχει παρουσιάσει. Κύριε Άοκεν. Ναι, δεν θέλω να εκφράσω τη θέση των πρασίνων, εκφράζω όμως τη θέση του Κοινοβουλίου ε, και της Επιτροπής και επανειλημμένος έχει αναφερθεί στις εκθέσεις μας και από τον ΟΗΕ. Όλος ο ΟΗΕ μιλά ξεκάθαρα για κατοχή. Είναι παράνομο. Ε, αυτό πρέπει να αναφερθεί κάπου. Πρόεδρος, θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο, στον κύριο Μπόσακ ο οποίος είναι ο διευθυντής της Ούνρα στην ε, Γάζα, στην κλωβά της Γάζας και με τηλεδιάσκεψη θα μας μιλήσει. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Um, it's a pleasure to be able to provide Σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να μπορούμε να παρουσιάσουμε μια σύντομη επισκόπηση για τις τελευταίες εξελίξεις. Την θέση αυτή ανέλαβα πριν από 10 ημέρες περίπου και μπόρεσα να επισκεφθώ ολόκληρη την περιοχή της Λωρίδας, της Γάζας. Είδα όχι μόνο την καταστροφή επικρατεί, αλλά και τις εντυπωσιακές προσπάθειες του τοπικού πληθυσμού να καθαρίσουν ε, τα συντρίμια και να υπερβούν τις προσπάθειες καταστροφής. Εμείς έχουμε ασχοληθεί με μικρές επισκευές και περιμένουμε να προχωρήσουν οι προσπάθειες ανοικοδόμησης των πλήρως καταστραμμένων κατοικιών. Έχουν ήδη φτάσει κάποια κονδύλια για την προσπάθεια νοικοδόμησης. Χρειάζονται όμως πολύ περισσότερα. Η μεγάλη, το μεγαλύτερο ποσό έρχεται από αραβικές χώρες και προς αυτούς στρέφεται ο πληθυσμός. Όμως πέραν της καταστροφής και της ανοικοδόμησης υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή η κατάσταση στην οποία ζει ο πληθυσμός εκεί. Βλέπουμε απελπισία και κραυγές ανθρώπων που αναρωτιούνται που να πάνε. Από τα σχολεία που επισκεφθήκαμε είναι εντυπωσιακό να παρατηρήσει κανείς ότι παρόλα αυτά ο κόσμος χαμογελάει. Υπάρχει διάθεση τα παιδιά να μάθουν, να μελετήσουν Θέλουν να εξαλειφθεί η βία και θα έλεγα ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να περάσει κανείς σε συζήτηση για το τι πραγματικότητα μπορεί να διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας για τους Παλαιστινίους. Παράλληλα όμως βλέπουμε και αυτό το λέω από την άποψη την αναπτυξιακή και την ανθρωπιστική, βλέπουμε ότι η κύρια μερίμνα του πληθυσμού αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τον αποκλεισμό, με τις συνέπειες στην καθημερινή του ζωή και επιπροσθέτως έχουμε και το θέμα με τα Αιγυπτιακά σύνορα. Έχουν πλημμυρίσει τα σύνορα Δεν θα περάσω σε σχόλια για τα θέματα ασφάλειας. Είδαμε δείγματα τελευταία από τη Λόριδα της Γάζας. Και όλοι είναι πολύ περισσότερο επικεντρωμένοι στις καθημερινές ανάγκες, στην επιβίωση. Το πρόβλημα είναι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που είναι συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες, η ποιότητα της, ε, των ε, καταστάσεων επεξεργασία των υδάτων, υπάρχει όλο ένα και περισσότερη ρήπανση, υπάρχει το θέμα της απασχόλησης, και το κατά πόσο μπορούν να πάνε για αλληλεία πέραν των 6-7 μιλίων που επιτρέπονται από την ακτή. Αυτές είναι καθημερινές ε, έγνοιες και επιθυμίες του πληθυσμού. Αυτές εκφράζει. Αυτό όμω που βλέπουμε να συζητιέται και ίσως και να είχε σημασία για την συζήτηση του τι κάνουμε εμείς εκεί σε συνεργασία με εσάς, είναι ότι βλέπουμε αυτές οι ανθρώπινες ανησυχίες συχνά να ε, μετατρέπονται σε μια πολιτική συζήτηση περί ασφάλειας. Εκεί με τους ε, πυράβλους ε, από τη Γάζα προς το Ισραήλ και τα αντίπινα τα κλασικά αντίπινα βλέπουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες αυτές τις επιθυμίες που εκφράζονται η συνολική εικόνα, το τοπίο που αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ως συνέπεια της όλης κατάστασης και της έκφρασης των αναγκών ασφάλειας επιτόπου φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των μελών της κοινότητας κίνδυνος για περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση. Υπάρχει και η διάσταση του λαθρεμπορίου, της παράνομης δράσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα που να μας επιτρέπει να τα ελέγχουμε αυτά με κατάλληλο τρόπο. Από τις συζητήσεις τις οποίες συμμετείχαμε τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε ότι όλοι στρέφονται προς την δική μας ομάδα εργασίας, ώστε να είμαστε ο βασικός πυλώνας σταθερότητα για να παράσχουμε κάποιες υπηρεσίες και πολύ μου λένε ότι στις δικές μας κλινικές έχουν γεννηθεί πολλοί από τους ε, ντόπιου. Ε, έχουν πάει σχολείο στα σχολεία μας, έχουν εμβολιαστεί στα νοσοκομεία μας. Είμαστε λοιπόν μακράν ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης. Περίπου 12 έως 13.000 Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας απασχολούνται από την Ούρα. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσει το μήνυμα στα μέλη της κοινότητας ότι πρέπει να συνεχίσουν να παράσχει αυτές τις βασικές υπηρεσίες που ε, ξεκινούν από τις ανθρωπιστικές ανάγκες και φτάνουν ως τα αναπτυξιακά και τα θέματα των δικαιωμάτων. Οπωσδήποτε Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να αποστείλουμε το μήνυμα προς τον πληθυσμό ότι είμαστε στο πλευρό τους και από την σκοπιά την ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή και ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτό το είδος τις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι ενώ πράγματι συνεχίζονται οι προσπάθειες ανεκοδόμησης, βλέπουμε αραβικές χώρες από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ να εμπλέκονται στην όλη προσπάθεια και λαμβάνουμε το μήνυμα ότι οι χώρες αυτές ε, εν μέρη μόνο συνεργάζονται μαζί μας περιορισμένα. Έχουμε ισχυρή στήριξη από τη γερμανική κυβέρνηση αλλά θέλουμε να ακολουθηθεί και η δέσμευση στο Κάιρο ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη για τις προσπάθειες ανεκοδόμησης της ΟΥΝΡΑ με τη συνεργασία φορέων και οργανισμών, τη συνεργασία του τοπικού πληθυσμού. Έχουμε 1,2-1,3 άτομα 1,2-1,3 εκατομμύρια άτομα που είναι πρόσφυγες σε αυτή την περιοχή. 500.000 δεν είναι. Πρέπει να ασχοληθούμε και με τις δικές τους ανάγκες και μίλησα και για τον παράνομο αποκλεισμό. Το εξετάζουμε και αυτό για να βεβαιωθούμε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας των σχολείων επιτυγχάνουμε το σκοπό, το σκοπό της και μπορούμε να παράσχουμε εκπαίδευση σε συνθήκες ουδετερότητας. Αυτό παραμένει μια κατεξοχήν προτεραιότητα για μας. Το έχω επισημάνει σε όλες τις συναντήσεις με τους υπευθύνους των σχολείων και κυρίως υπάρχουν πολύ στρατευμένες νεαρές γυναίκες που συμμερίζονται αυτό τον σκοπό, αποφασισμένοι νέοι που θέλουν τα πράγματα να αλλάξουν και να πάρουν μια τροπή ειρηνική. Θέλουν να μελετήσουν, να σπουδάσουν και να βρουν δουλειά. Όπως και τόσοι άλλοι. Όσο αφορά τα ζητήματα προστασίας των παιδιών, βλέπουμε διαφορετικές ε, εκθέσεις να συγκεντρώνουν στοιχεία για το θέμα αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά από συνέπειε λόγω των σειράξεων και είναι τραγικέ οι συνθήκε στις οποίε ζουν τουλάχιστον 500 παιδιά λόγω της όλης κατάστασης. Κοιτάζουμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε εσωτερικώς για την αντιμετώπιση κρίσεων από την άποψη ετοιμότητας περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων και ούτω καθεξής. Πάντως το βασικό μήνυμα που λαμβάνω από τον πληθυσμό είναι ότι αυτό που θέλουν εκείνοι να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τις βασικές δραστηριότητες που έχουμε ήδη ξεκινήσει, δηλαδή εκπαίδευση, υγειονομικές υπηρεσίες και να συνεχίσουμε να είμαστε ένας πυλώνας σταθερότητας σε αυτή τη θάλασσα, την ταραγμένη. Αυτό θα πει ότι και εργασία θέλουν να συνεχίσουμε να προσφέρουμε για να έχουν κάποια προοπτική και για το μέλλον. Και η αναπτυξιακή διάσταση από ανθρωπιστική σκοπιά είναι αυτό που τους απασχολεί κάπως λιγότερο. Αυτό που θέλουν είναι να έχουν μια εξωπρεπή ζωή, να είναι υπερήφανοι για όσα κάνουν και να ζουν μια ζωή όπου μπορούν να στηρίξουν, να επιτρέψουν στις οικογένειές τους να επιβιώσουν. Σας ευχαριστώ για την επαφή αυτή, την ε, δουλειά που σας είπα αυτή την ανέλαβα εδώ και δέκα μέρες μόνον. Είμαι λοιπόν στο να έχουμε διάλογο και συζητήσεις και θα είμαι πρόθυμος στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ρόκο Πολίν για την Παλαιστίνη και τον Νίκο Χριστοφόρου για το Ισραήλ, αν με έχουν ενημερώσει. Καλά. Παρακαλώ. Βεβαίως, με τον συνάδελφο Νίκο από, για το Ισραήλ και την Πέτρα για την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή θα σας ενημερώσουμε. Ουσιαστικά ήρθαμε για να ακούσουμε ε, τις δικές σας αναφορές, θα διαβάσουμε και τις εκθέσεις. Σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προωθεί τις ανησυχίες που έχουμε και τις γνωστοποιεί στους εταίρους μας από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Ευχαριστούμε και την Ούνερα για την ανεκτήμητη δουλειά που κάνουν σε όλα τα πεδία, αλλά κυρίως στη Λοίδα της Γάζας. Θα ήθελα τώρα σε σχέση με τα ευρήματα της αποστολής να σας ενημερώσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 100% των πλέντιστρων από το Κάιρο και το 70% ήδη έχει ε, εκταμιευτεί. Φυσικά ε, ε, για την ενέργεια και το, την ενέργεια συγγνώμη, και το πόσιμο νερό είναι κέρια σημασία και προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Προσπαθούμε να βρούμε και επιπρόσθετα κονδύλια πέρα από αυτά τα πλέντε, πέρα από τις δεσμεύσει που έχουμε και θα έχουμε νέα τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Θα ήθελα κλείνοντας να σας ευχαριστήσω και πάλι για την επίσκεψη που κάνατε και για το follow-up είμαστε στη διάθεσή σας ε, και για οποιοδήποτε θέμα μπορούμε να συνεργαστούμε. Πολύ ωραία. Για την Ισραήλ, ο Νίκος Χριστοφόρου, παρακαλώ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ωραία. Ε, ο εκπρόσωπος από την πρεσβεία του ή εκπρόσωπος από την πρεσβεία του Ισραήλ είναι εδώ. Θέλετε το λόγο. Ο Ρίτσαρτ Χάουιτ νομίζω έχει μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Μπορείτε να με ακούσετε. Θέλω να απευθύνω την ερώτησή μου στον ε, διευθυντή της Ούνρα. Ε, Βέβαια σας ακούω. Σύντομα θα μιλήσω, διότι σίγουρα δεν έχετε χρόνο, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία για μας ε, να μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ανταλλαγή με απόψεων με εσάς μετά το διορισμό σας και από ό,τι ξέρω και από τους δύο προκατόχους σας είναι ε, πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος σας για την ελευθερική διαδικασία και για τη Γάζα όλος ιδιαίτερος. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Θα ήθελα μόνο να πω ότι από πλευρά του Κοινοβουλίου είμαστε περήφανοι και υποστηρίζουμε την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει επιπρόσθετα κονδύλια που υποσχέθηκε τον Αύγουστο, διότι χρειαζόμαστε αυτά τα κονδύλια για να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία στη Γάζα και υποστηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια. Είμαστε περήφανοι επίσης διότι σας υποστηρίζουμε ε, στο έργο σας. Ε, είμαστε σταθεροί εταίροι και ε, παρέχουμε και εμείς βοήθεια. Είστε πολιτικά ουδέτεροι, υποστηρίζετε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την επίλυση της διένεξης και με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτό που είπατε για τα σχολεία στη Λωρίδα της Γάζας. Τι? Ε, τα, για το, και τα, τα μαθήματα που γίνονται για το ολοκαύτωμα και θα πρέπει να προβληθεί ε, το έργο σας ε, και ούτω άλλω μα ενημερώνετε για μας θα ήταν πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε την κατάσταση αν δεν ήσασταν εσεί επιτόπου. Ε, και ε, ως πρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας για τη Μέση Ανατολή εδώ στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω να έρθετε να μας δείτε όταν έρθετε στην Ευρώπη για να κάνουμε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, να πω κλείνοντας, ε, έχει ε, ιδιαίτερο ειδικό βάρος όταν μιλάμε για τα εγκλήματα πολέμου στη Λόριδα της Γάλλης στο παρελθόν, είτε μιλάμε για την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, είτε μιλάμε για το ανθρωπιστικό διάδρομο από την Κύπρο προς τη Γάζα, έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος το ανθρωπιστικό δίκαιο. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό και είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχω την ευκαιρία να το πω σήμερα. Καλή επιτυχία και πάλι και θα κλείσω εδώ. Ο Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Το πρώτο είναι το εξή. Η Ούνρα ε, απασχολεί 12 με 13.000 Παλαιστινίους. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ουδετερότητα. Όταν είναι τόσοι πολλοί Παλαιστίνοι οι οποίοι απασχολούνται από την Ούνρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της είναι αυτές που έχουν δώσει ένα μεγάλο μέρος των 2,6 δισεκατομμύριων που έχουν μπει στην ε, περιοχή αυτή. Αυτή είναι μια σημαντική υποστήριξη βέβαια. Ποια είναι η πιθανότητα οι αραβικές χώρες να μπορέσουν να δώσουν μεγαλύτερη χρηματική συνεισφορά. Κάτι το οποίο είναι προς το συμφέρον τους. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που θέλετε να διατυπώσετε για τον κύριο Σάκ. Εάν όχι, του δίνω αμέσω το λόγο για να απαντήσει εν συντομία στο ερώτημα που ετέθη από τον κύριο Γκέργε και από τον κύριο Χάουτ φυσικά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Σάκ. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για, την, για τα θερμά σας λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν για την συζήτηση αυτή και φυσικά για τη δυνατότητα σε μια μεταγενέστερη στιγμή να έχω περισσότερες συζητήσεις με την Επιτροπή σας. Έρχομαι στο θέμα της υποστήριξης από τις αραβικές χώρες. Είναι φυσικά ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε κι εμείς. Το θέμα της ευρύτερης υποστήριξης που μπορεί να δοθεί στη Γάζα. Αλλά με την κάπως περιορισμένη γνώση που έχουμε αυτή τη στιγμή η προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας, το μήνυμα που πήραμε σχετικά με την ανοικοδόμηση αυτή, είναι ε, ότι οι αραβικές χώρες είναι αυτές που ηγούνται τις προσπάθειες ανοικοδόμησης, είναι οι κύριοι χορηγοί για την ανοικοδόμηση της Λόριδας της Γάζας και λένε ότι θα θέλανε να υπάρξει μια μεγαλύτερη υποστήριξη και μεγαλύτερη εφαρμογή σχεδίων από τις άλλες χώρες και οντότητες που υποστηρίζουν αυτήν την ε, διαδικασία ανοικοδόμησης. Προς το παρόν μόνο η Γερμανία υποστηρίζει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης. Αυτό φυσικά εμποδίζει κάπως την δυνατότητά μας να παροτρύνουμε τους Άραβες τα αραβικά κράτη σε μεγαλύτερη συνεισφορά για τα θέματα αυτά. Επίσης, θέλω να πω ότι αναγνωρίζω τη σημασία της ε, προσπάθειας μαζί με τους μαθητές να προωθήσουμε μηνύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μηνύματα συμφιλίωσης με την Ισραηλινή πλευρά. Συμφωνώ απόλυτα με κάτι τέτοιο, απλώς τονίζω ότι αυτό που βλέπω όλο και περισσότερο στα μάτια των παιδιών που συναντώ είναι ότι θέλουν να μάθουν για να μπορούν να έχουν δουλειά όταν μεγαλώσουν. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σε επίπεδο ανθρώπινο, σε επίπεδο ανάπτυξης, είναι να προωθήσουμε όλο και όσο είναι δυνατόν μια κατάσταση πραγμάτων όπου η ελκυστικότητα των ριζοσπαστικών λύσεων είναι λιγότερη από ότι το να προσπαθήσει κανείς να έχει μια φυσιολογική ζωή. Έχουμε δει βέβαια ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με την εκτόξευση πυράβλων από την ε, πλευρά της ε, Γάζας και γνωστή απάντηση από την πλευρά του Ισραήλ, αλλά είδα πάρα πολλά αποφασισμένα πρόσωπα, πάρα πολλά παιδιά τα οποία χαμογελούν και πηγαίνουν στο σχολείο και συνεχίζουν την προσπάθειά τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάκ. Για τις απαντήσεις που μας δώσατε τώρα για να κλείσουμε τη συζήτηση, μήπως θέλει ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ να προσθέσει κάτι. Διηγηθήκατε της αντιπροσωπείας. Όχι, ωραία. Θα περάσουμε στο σημείο 5 της μέσης διάταξης. Είναι η έκθεση της Υποεπιτροπής ε, για την Ουκρανία. Ο Ρίτσαρτ Χάουιτ ε, ήταν ο πρόεδρος σε αυτή την αποστολή. 21-24 Ιουλίου πήγατε στην Ουκρανία. Ο στόχος ήταν να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση προς τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τις προκλήσεις που συνδέονται με εσωτερικά εκτοπισμένους ε, τις λύσεις ενδεχομένως για την ε, σύγκρουση για την κατάσταση που προέκυψε από την παράνομη προσάρτησή της Κρυμαίας ε, καθώς και τη νομοθετική προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση ε, στο δεύτερο τμήμα της αποστολής ε, μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων συζήτησαν αυτό το ζήτημα σε συνεδριάσεις σε υψηλού επίπεδου την έκθεση που πραγματικά θα τη λάβουν οι βουλευτές να αναφέρω ότι ο πρόεδρος αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου με την Ουκρανία, το Αντρέ Πλένκοβιτς, ε, είναι εδώ πέρα. Θα ακούσουμε τον Ρίτσαρτ Χάουι τώρα. Ρίτσαρτ, ε, έχεις το λόγο. Άλλη μια περιοχή με συγκρούσεις όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα σαφώς παραβιάζονται δύσκολο σε αυτή την Επιτροπή να αποδώσουμε τη σημασία που πρέπει σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αλλά το προσπαθούμε. Πέντε μέλη της Επιτροπής μας επισκέφθηκαν την Ουκρανία, ενωθήκαμε με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το τελευταίο τμήμα της αποστολής μας. Ήταν πολύ αποτελεσματική αυτή η συνένωση. Από τη δική μας Επιτροπή ο κ. Ντεμεσμάκερ, ο κύριος ε, από τους φιλελεύθερους και όπως είπατε ο κύριος Πλένκοβιτς επικεφαλής αντιπροσωπείας αλλά και εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες και να ευχαριστήσω και τη γραμματεία από καρδιάς. Ευχαριστούμε για όλη σας τη στήριξη και το προσωπικό της ομάδας που μας στήριξαν. Τα απορίσματα τώρα της έκθεσης. Ασχοληθήκαμε με θέματα ελευθερίας της κυκλοφορίας και μεταχείρισης των προσφύγων, ιδίως σε σχέση με τους εσωτερικούς μετατοπισμένους, καθώς η Ουκρανία ξεφεύγει από την κρίση. Να καταστήσω σαφές ότι και σε αυτή την έκθεση και στα σχόλιά μου Σκοπό δεν έχω να ανοίξω μια δεύτερη συζήτηση για, την πολιτικές, για τα πολιτικά πράγματα στην κρίση της Ουκρανίας. Έχουμε όλες τις δικές μας ε, σκέψεις. Το γεγονός ότι επικεντρωθήκαμε στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επικριτική στάση προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Πολλοί από εμά είμαστε θετικά διακείμενοι προ αυτή την κυβέρνηση Ήθελαμε να δούμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πόσο γρήγορα μπορέσαν να προστατευτούν και πόσο έγιναν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα από όλου του φορεί ε, στην Ουκρανία. Βρήκαμε παραβιάσεις στην περίπτωση του 1 εκατομμυρίου εξωτερικών εκτοπισμένων σε διάφορε περιοχέ και ιδίω στην Κρυμαία. Υπάρχουν σοβαρέ μέρημνε για την ε, πρόσβαση, την ανθρωπιστική πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές, για την ελεύθερη κυκλοφορία των οικογενειών που θέλουν να συνενωθούν ξανά και για την σωστή καταγραφή του καθεστώτος πρόσφυγα. Με συγχωρείτε, αλλά αν θα θέλατε να ε, Θέλαμε λοιπόν να δούμε αν μπορούν οι πρόσφυγε να καταγραφούν σωστά και να λάβουν τη στήριξη που του αξίζει ω προ την ελευθερία κυκλοφορία. Κατέστη σαφέ ότι ενώ υπάρχουν ανησυχίε ασφαλεία από την ε, κυβέρνηση της Ουκρανίας και εσωτερικώ υπάρχουν απειλέ για τρομοκρατικέ επιθέσει. Υπήρχαν επίση και μέρημνε για τον περιορισμό τη ελευθερία κυκλοφορία. Δηλαδή κάποιοι αναγκάζονται να φύγουν ε, μέσα από περιοχές που υπάρχουν άρκες και απειλούνται οι ζήτους. Επίσης, Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν προσφέρεται η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει διατεθεί από επίσημους φορεί του ΟΗΕ. Όμω είχαμε επικοδομητικέ συζητήσει με του Ουκρανού εταίρου για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ιδίω. την ε, συστηματική δωροδοκία ορισμένων και τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν σχετικά για να λάβουν βοήθεια από τους κυβερνητικούς φορείς να ε, σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση. Επίσης, συναντήσαμε εκπροσώπους από την Κρυμαία οι οποίοι μας ζητούν, ζητούν από το κοινοβούλιο μας να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Κρυμαία με όλα τα θέματα της ελευθερίας της κυκλοφορίας, τα οποία ακόμη απασχολούν. Δεν μιλάμε για τις περιοχές όπου υπάρχουν ε, συγκρούσεις ή αναταραχή, αλλά ιδιαίτερα για την Κρυμαία. Συζητήσαμε με την ε, κρίση που μπορεί να έχει της κατάστασης στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την κατάσταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και τις περίπτωσες παρανομίας ή όχι, αλλά η αργή κύρωση είναι ένα κάπως ανησυχητικό θέμα. Ελπίζουμε ότι όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό μήνυμα που λάβαμε. Αλλά πρέπει να πιέσουμε οι διώξεις για τις υποθέσεις της πλατείας Μαϊντάν είναι επίσης ένα θετικό δείγμα. Θα σχηματιστεί ανακριτική επιτροπή γι' αυτό, αλλά ακόμη δεν είδαμε να υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία ότι η εισαγγελία προχωρά γρήγορα. Θα πρέπει να κινηθεί και τα θύματα να δικαιωθούν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάθε διπλωματική προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Επίσης ασχοληθήκαμε με το θέμα της ανταλλαγής ε, φυλακισμένων, κρατουμένων. Ίσως κρατούμενοι δεν είναι ο σωστός όρος, γιατί και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης κάποιοι έχουν συλληφθεί και κρατούνται ίσως και μυστικός και οι δύο πλευρές ξέρουν ότι η άλλη πλευρά τους έχει ε, σε κράτηση ε, νομίζουμε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ρυθμού Σταυρού είχε πρόσβαση και οι διαπραγματεύσεις για τις ανταλλαγές κρατουμένων υπονοούν ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση σχετικά. Όμως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όσοι κρατούνται παρανόμως ή ανωνύμως μπορεί να υποβάλλονται σε στερήσεις ή άλλες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε ή να αντιληφθούμε ποιοι κρατούνται, πού και να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια που μπορεί να καταβάλλεται ώστε να γίνουν ε, οι ανταλλαγές κρατουμένων. Επίσης για τη διαφθορά και τη διαφάνεια ακούσαμε σχετικά στοιχεία, δεν θα πω πολλά για αυτά. Πάντως η αντιπροσωπεία εντυπωσιάστηκε από τις Ουκρανικές αρχές για την, για την προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με τεράστια φαινόμενα διαφθοράς και φαίνεται να υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για να αναχαιτιστεί η κατάσταση αυτή. Ε, με τις ε, με την ε, στάση της Ευρώπης που προσπαθεί να βοηθήσει. και παρά τις αντιστάσεις ε, της δεξιάς πτέρυγας ή τις αναταραχές που προσπαθούν να προκαλέσουν. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχει αυθεντική επιθυμία από την Ουκρανική κυβέρνηση να αφοπλίσει τις ομάδες που είναι επιθετικές και να διασφαλίσει τα δικαιώματα όλων των πολιτών και το δημοκρατικό πολιτεύμα της χώρας. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Ένα, ότι τα ότι διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα οργανώθηκε την ίδια εβδομάδα που ήμασταν εκεί, οπότε είχαμε και ένα κοινοβουλευτικό σκέλος στις συζητήσεις μας. μπορέσαμε να συζητήσουμε με κυβερνητικούς εκπροσώπους και να θέσουμε το θέμα σε όλη του τη σημασία. Κάποιοι ανησυχούν με την ε, βαρύτητα της κρίσης που συνεχίζεται στην Ουκρανία. Και φαίνεται να μην είναι η πρώτη πολιτική προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμω εμεί θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή προτεραιότητα, διότι αυτό ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε στι σχέσει μα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία. Τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν ουσιαστικέ οι προσπάθειέ μα να χτίσουμε το δημοκρατικό πολιτεύμα, να στηρίξουμε τον δημοκρατισμό σε αυτή τη χώρα και είναι μεγάλη μα χαρά να στηρίζουμε τι σχετικέ προσπάθειε. Τέλο, για του συναδέλφου που βρίσκονται στην αίθουσα και γενικώ στο κοινοβούλιο, καθένα εδώ μιλά για πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τους πρόσφυγες της Συρίας και το συζητάμε γιατί ξαφνικά μιλάμε για μια μείζωνα πολιτική κρίση στην Ευρώπη, οπότε έχει λάβει πολιτική προσοχή. Όμως να μην μιλάμε μόνο για την τρέχουσα κρίση, για την πρόσφατη κρίση. Υπάρχουν και άλλες εξέλιξεις Ήρθαμε από την Ουκρανία έχοντας την αίσθηση ότι η σύγκρουση δυστυχώς διαρκεί όπως και πριν υπάρχουν παραβιάσεις στην εκεχηρία και δυστυχώς αυξάνονται και δεν μειώνονται και οι ομάδες των επαναστατών έχουν ξαναρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους. Είναι πολλά τα στοιχεία για πρόσφυγες που μακροπρόθεσμα δεν έχουν κάποιο καθεστώς που να τους προστατεύει, λύσεις που να τους ε, καθησυχάζουν και η κυβέρνηση ανησυχεί από τα δείγματα που λαμβάνει από τον πληθυσμό που ε, ε που παίρνει ε, την κατεύθυνση της φυγής ή τέλος πάντων δεν έχουν ακόμη τα οικονομικά μέσα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώνεται στην Ουκρανία και πιστεύω ότι η αποστολή μας ε, και άλλες σχετικές προσπάθειες θα μπορέσουν να ανακαιχθήσουν αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε κύριε Χαούτε, Κύριος Πλένκοβιτς τώρα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βαλενσιάνα. Εφόσον έχουμε διερμηνείς θα μιλήσω κροατικά. Πρώτα απ' όλα με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα σε αυτήν την μεικτή αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής ΔΡΟΑ για την Ουκρανία. Είναι η ένατη φορά ε, τον περασμένο χρόνο που επισκέπτομαι την Ουκρανία. Και το θετικότερο για τα μέλη της Επιτροπής είναι να συνειδητοποιήσουμε με ποιο τρόπο δραστηριοποιούνται τα διάφορα θεσμικά όργανα της Ένωσης επί τόπου. Η Επιτροπή Επιτροπή Άμυνα, η Επιτροπή Προπολογισμών, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετέβησαν ήδη στην Ουκρανία και μην ξεχνάμε πω η Επιτροπή Εμπορίου και άλλε επιτροπέ θα επισκεφθούν την Ουκρανία πέρυσι. Συμμετείχαν και οι φίλοι μας από την Ουκρανία, έχουμε μια ομάδα φίλων, έχουμε ειδικό εισηγητή, είναι ευρύτατο το φάσμα των δραστηριοτήτων και αυτό δείχνει πόσο σημαντικός εταίρος είναι για μας η Ουκρανία. Θα ήθελα να σχολιάσω την τελευταία πρόταση του κυρίου Χάουιτ. Μίλησε για την ανθρωπιστική κρίση που ακολουθεί διαφορετικούς δρόμους ακόμη και την Κροατία. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουμε στην Ουκρανία και σχεδόν 1 εκατομμύριο έχουν ήδη φύγει ε, κατευθυνόμενοι προς τη Ρωσία και άλλες χώρες. Η κρίση στην Ουκρανία είναι πολύ διάστατη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις διαστάσεις και, τους, ε, και τα πολλά και διαφορετικά μέρη της ε, διένεξης. Η Ουκρανία πάντως έχει αναλάβει σοβαρή δέσμευση για την υποστήριξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποστολή μεταξύ άλλων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στον Τονέτσε και στο Λουκάνς να παρακολουθεί την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στην Κρυμαία που προσαρτήθηκε παράνομα. συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα και αποφασίσαμε να διοργανώσουμε και μια ακρόαση για να ακούσουμε και τα μέλη των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ανθρωπιστικών οργανώσεων που ε, δραστηριοποιούνται επί τόπου. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να παραμείνει η προτεραιότητα αυτό το ζήτημα. Ε, ε εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών της ε, Ουκρανίας. Στη συνεδρίασή μας ε, τον Ιούλιο υποστηρίξαμε την ιδέα να δοθεί το δικαίωμα και στους πρόσφυγες να ψηφίσουν θα πρέπει να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν παρότι έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από τον τόπο διαμονής τους, ε, κάτι που ούτως ή ε, δεν έχουν επιλέξει οι ίδιοι, παρά λοιπόν την απόσταση από τον τόπο διαμονής τους ε, πρέπει να φροντίσουμε να ψηφίσουν. Οι αρχές στα κατεχόμενα προσπαθούν να διοργανώσουν εκλογές ε, που αντίκειται στην ε, ε, κείμενη νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο θα στείλει 7 παρατηρητές για την εκλογική διαδικασία και φυσικά εάν δεν διεξαχθούν οι εκλογές βάσει της νομοθεσίας δεν μπορέσουμε εμείς να αναγνωρίσουμε ως έγκυρα τα αποτελέσματα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι υπάρχουν και σχετικές ε, απαιτήσει από τη Συμφωνία του Μίνσκ. Ε, μέσα από τέτοιες ε, δράσεις μπορούμε να είμαστε σε διαρκή επαφή με τους εκπροσώπους της κοινωνίας της Ουκρανίας. Επισκεφθήκαμε επίσης να σας πω ε, καταβλισμούς προσφύγων ε, και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για τις ανάγκες τους. Οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ο κύριος Στυλιανίδης, στην Επιτροπή και συνάδελφοι από διάφορες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από άλλα θεσμικά όργανα που συνεργάζονται ε, με την ε, υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ε, και οι δικές τους προσπάθειες είναι πάρα πολύ σημαντικές διότι φροντίζουν τα παιδιά, τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους Ξέρω ότι κάποιος άλλος συνάδελφος θα ασχοληθεί όλος ιδιαίτερος με το ζήτημα, δηλαδή για την προστασία των ε, παιδιών αύριο στο Κοινοβούλιο. Ήταν πολύ επίκαιρη η επίσκεψή μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος ε, με την Ουκρανία με τη συμβολή της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πλένκοβιτς. Ξέρουμε ότι θα συνεχίσετε να συνεργάζεστε με την αρμόδια, με την αντιπροσωπεία και την Επιτροπή μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουκρανία. Ο κύριος Τέμες Μάκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, δεν σας εκπλήσει πάρα πολύ αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Χάουιτ που ηγήθηκε τη αντιπροσωπία ε, και να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπου συναδέλφους που ήρθαν στην Ουκρανία. Τους ευχαριστώ για την εξαιρετική αυτή συνεργασία που είχαμε. Ήταν πολύ καλή, πολύ επιτυχημένη η αντιπροσωπεία. Ε, είναι πολλά τα δάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν την επίσκεψη και κάναμε και μια συνεδρίαση ε, στην αντιπροσωπεία μας, ε, στην ομάδα δηλαδή ε, διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και Ταυτόχρονα έκανα και κάποιες ε, έρευνες ε, για επιμέρους ζητήματα όπως η ελευθερία μετακίνησης ε, στην Ουκρανία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διότι εμποδίζονται άνθρωποι, δεν έχουν την, πλέον αυτή την ελευθερία μετακίνησης, δεν μπορούν να επισκεφθούν την οικογένειά τους, τους φίλους τους που διαβιούν από την άλλη πλευρά της γραμμής διαχωριστικής γραμμής. Υπάρχουν τα προβλήματα διαφθοράς. Η ηλεκτρονική καταγραφή λειτουργεί καλά. Στην αρχή υπήρξαν κρούσματα παιδικών ασθενειών, αλλά άμα δείτε το, την ιστοσελίδα θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ φιλική προς το χρήστη και μπορεί εύκολα κάποιος ε, να κάνει την εγγραφή και μετά την εγγραφή σε αυτούς τους καταλόγους μπορεί να διασχίσει την διαχωριστική γραμμή ε, και να περάσει από την άλλη πλευρά. Συγχαίρουμε την Ουκρανική κυβέρνηση. Στη συνέχεια, ο κ. Πιμκίν, ε, με τον οποίο συναντηθήκαμε στο Κίεβο, μας ε, μίλησε για τα κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας ε, κατά μήκο ε, της γραμμής. Τώρα το Σεπτέμβριο άρχισε να λειτουργεί το κέντρο στο Αρτιμόσκ κατά μήκο της διαχωριστικής γραμμής υπάρχει μία αλυσίδα λογιστικής επιμελητίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και μπορούν όλοι να αγοράζουν εκεί φάρμακα, ε, τροφή σε προσιτές τιμές, ε, μπορούν ε, να σηκώσουν χρήματα από το λογαριασμό τους. να κάνουν τις διοικητικές διατυπώσεις που πρέπει να κάνουν. και η προσέλευση είναι περίπου 5.000 ε, άνθρωποι την ε, ημέρα. Τέτοια κέντρα λογιστικής επιμελητίας ε, θα λειτουργήσουν κατά μήκο της διαχειριστικής γραμμής. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά πολύ θετική αυτή η εξέλιξη. Φυσικά δεν ελέγχουμε καθόλου τα κατεχόμενα εδάφη, Ντονιέτς και Λουγάνσκ, οι διάφορες ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, κάνουν θλιβερές αναφορές, ε, δεν υπάρχει κανένα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην φλαμανική τηλεόραση είδα έναν, την αναφορά από έναν Ολλανδικό, ε, Ολλανδό συγγνώμη, δημοσιογράφο που χρόνια εργαζόταν στη Ρωσία και που πήγε επανειλημμένα στα κατεχόμενα και είπε πως είναι σοβαρότατη κατάσταση και είναι πολύ κακή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, έχει καταληθεί και ε, υπάρχουν ε, λήψεις ε, τροφίμων, φαρμάκων, είναι διαθέσιμο μόνο σε εξωφρενικές τιμές και μια οργάνωση τύπου Κάριτας μας έδωσε μια ζωφερή εικόνα της κατάστασης. Λάβαμε επίσης και με email την έκθεση της ΟΝΤΡΙ του SRM για τη, τις αρμοσίες δηλαδή για τις εθνικές μειονότητες και ε, της ε, ε, οργάνωσης για τους δημοκρατικούς θεσμούς και πρόκειται για την Κρυμαία εκεί. Είναι μια εκατοστή σελίδες τη έκθεσης και βλέπουμε την εικόνα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι, ε, επιδεινώνεται διαρκώς ε, η ήδη πολύ κακή κατάσταση. Δυστυχώς ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε πίεση στην Ουκρανική κυβέρνηση και μετά το Μέντεν υπάρχει καλή βούληση αλλά δεν μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στη, στο, στους Ρώσους. Οι Ταρτάροι στην Κρυμαία και ε, η κατάσταση των μειονοτήτων, η ελευθεροτυπία, συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Έχουν μπλοκάρει τους δρόμους πρόσβασης που είχαν παραμείνει ανοιχτοί, Η Κρυμαία, όπως και να το κάνουμε, εξαρτάται από την Ουκρανία για την τροφοδοσία. Τώρα λοιπόν έχουν αρχίσει να κλείνουν και τους δρόμους για να μπορέσουν να τραβήξουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας ε, σε αυτό που τους συμβαίνει. Θα σταματήσω εδώ. Ε, είναι εξαιρετικός ο διάλογος που είχαμε με την Ουκρανία για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά και η οικονομική κατάσταση είναι δεινή. 11% επιβράδυνση της ε, οικονομίας ε, στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε ότι 1,5 ε, εκατομμύρια άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Ουκρανία. Υπάρχουν αποκλεισμένες περιοχές. Εδώ συζητήσαμε ε, συζητάμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο κατανομής 160.000 ε, προσφύγων. Καταλαβαίνετε την τάξη μεγέθους. Εκεί είναι 1,5 το εκατομμύριο οι πρόσφυγες και πρέπει κάπου να στεγαστούν και κάπου να... Ε, διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι και ε, τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να παράσουμε πρακτική ε, υποστήριξη στην ε, Ουκρανία. Το ΜΕΝΤΑΝ ε, ήταν ένα κίνημα της κοινωνίας των πολιτών και ο στόχος ήταν να οικοδομήσουμε μια νέα Ουκρανία επί βάση των σύγχρονων ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών. Και τι έγινε, δέχτηκαν επίθεση από την γειτονική χώρα εξαιτία αυτού με όλες τις συνέπειες και σε επιπτώσεις που ξέρουμε είναι καθήκον μας να τους βοηθήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ζητάμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην δική μας υποεπιτροπή και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να παραμείνει ε, προτεραιότητα το ζήτημα της Ουκρανίας. Η κοινωνία των πολιτών, και θα κλείσω εδώ, ε, είναι εξαιρετικά δραστήρια. Είναι ισχυρή η δέσμευσή της για την υποστήριξη των δημοκρατικών αξιών και στο Λουγάνξε και στον Τονές πολλοί εθελοντές μοίραζαν φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα των εσωτερικά εκτοπιστέντων στην διαχωριστική γραμμή ε, ε, έφεραν, ε, έφεραν ε, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τα ρούχα για αυτούς τους ανθρώπους. Ε, πραγματικά ε, θαυμάζουμε την Ουκρανική κυβέρνηση και τις προσπάθειες που κάνει καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Ο κύριος Σωστορίτσιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επίκαιρη η επίσκεψή μας. Μπορέσαμε να ε, να δούμε, όπως είπε και ο κύριος Χάουιτ, πολλά πράγματα και θέλω να εξάρω τις ε, προσπάθειες του κυρίου Χάουιτ και την οργάνωση αυτής της αποστολής. Είχα μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων από την ευρωπαϊκή πλευρά με τους Ουκρανούς συνομιλητές μας και στο Νιεπρο, και στο Κίεβο. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη ε, επιτυχία η αποστολή μας γιατί ήταν αποστολή με συνεργασία και όχι με επικάλυψη προσπαθειών. Πήγαμε στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας και φέραμε το μήνυμα αυτό σε όλους τους συνομιλητές μας για, το, για αυτούς που είδαμε, σε αυτούς που είδαμε στο Κίεβο στη συνέχεια για την κατάσταση εκεί. Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία δεν είναι μονάχα δύσκολη κοινωνικά και οικονομικά. προς το παρόν μια σύνταξη στην περιοχή αυτή είναι περίπου 60, κάτω από 60 ε, ευρώ και ένας μέσος μισθός στο Κίεβο τώρα είναι, είναι περίπου 200 ευρώ. <clears throat> αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση σε οικονομικό επίπεδο σε αυτή την τόσο αχανή και οικονομικά πεπλεγμένη χώρα. Παρόλα αυτά. είδα να υπάρχουν μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται από τις τοπικές και τις εθνικές αρχές για να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση. Γενικά <clears throat> πιστεύω ότι η Ουκρανία είναι σε μια φάση οικοδόμησης και όχι απεικοδόμησης. Παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, βλέπουμε κάθε μέρα να έχουμε εκθέσεις για νεκρούς και τραυματισμένους στα ανατολικά σύνορα και υπάρχει τεράστια οικονομική κάμψη λόγω της προσάρτησης ε, εδαφών που ήταν στο παρελθόν τα κύρια και μάλλον και την, τον πόλεμο σε εδάφη που ήταν πριν η κύρια ατμομηχανή ανάπτυξης της ε, Ουκρανίας ιδίως σε βιομηχανικό επίπεδο αλλά πρόσφατα μαζί με τον συνάδελφό μου τον κύριο Κέρσμαχερ ήμασταν στην ε, λεγόμενη συνδιάσκεψη ΓΕΣ, συνεργασίες δηλαδή Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε τα πάνελ. Τα πάνελ είχαν πολλούς ε, από την κυβέρνηση που γυαλίζει το μάτι τους και έχουν μια τεράστια αφοσίωση στο έργο τους. Έχουν ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλη γραφειοκρατία και πολύ διαφθορά. Αλλά αυτοί είναι οι νέοι άνθρωποι που είναι οι υπουργοί και ανώτατα στελέχη σε διάφορους φορείς νομίζω ότι θα φέρουν μεγάλη αισιοδοξία και αυτή τη χρειαζόμαστε και εμείς για να δούμε αυτή την χώρα να προχωράει προς τα εμπρός. Η κίνηση των προσφύγων είναι σημαντική, είναι μεγάλη και έχει μεγάλο αντίκτυπο στα κεντρικά και τα ανατολικά τμήματα της χώρας, το προσφυγικό ρεύμα και οι συνθήκες τις οποίες υποδέχονται τους πρόσφυγες αυτούς είναι προς το παρόν ιδιαίτερα πρωτόγονες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να επιβιώσουν σε σχεδόν άδεια δωμάτια. Επισκεφτήκαμε και το είδαμε με τα μάτια μας. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αισιοδοξία και είναι καταπληκτικό πως οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Και πάλι θέλω να υπογραμμίσω το ότι είναι πολλές και καλά οργανωμένες ΜΚΟ που εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συναντήσαμε πάρα πολλούς. Δεν μπορούσα εγώ να μετρήσω πόσοι ήταν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ που μπορέσαμε να συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο και στο Κίεβο. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι το εξή ότι έχουμε πρόσβαση σε ανεξάρτητη και αμερόληπτη πληροφόρηση που μπορούμε να την συγκρίνουμε με τα στοιχεία που μας δίνει η κυβέρνηση. Τα άτομα αυτά, οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ, μιλάνε ανοιχτά για τη διαδικασία ανεξελίξη και μας δίνουν καλύτερες και όλο καλύτερες εκθέσεις για τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτές τις ΜΚΟ, να τις προσκαλέσουμε στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε την άποψή τους, για να συνεχίσουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους. Μας δόθηκε μεγάλη βοήθεια και από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κύριο Γιάννη και την ομάδα του που έχουν φέρει σε, πολύ, σε πέρα σε ψηλό επίπεδο την αποστολή τους και ελπίζω ότι θα παραμείνει η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αναβαθμιστεί τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν τις ακροάσεις μας <clears throat> για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία. Ήταν πολύ θετική η απόφασή μας να συγκεντρώσουμε και να συμπηλήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να ε, δημιουργήσουμε μια δική μας έκταση για την κατάσταση στην Ουκρανία. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να δείξει την ε, προσήλωσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά οι πληροφορίες που μας δίνουν οι ΜΚΟ θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτή την έκθεση υψηλού επίπεδου. Τέλος. Επειδή η κατάσταση δεν δείχνει σημεία βελτίωσης, ο χειμώνας που έρχεται θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις και δυσκολίες. Θα γίνουν πιο δύσκολες οι δυσκολίες που έχουμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συλλογής ρούχων και θα υπάρχουν και κοντέρνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα τοποθετηθούν να φέρουμε για να συλλεχθούν ρούχα και άλλα αγαθά για τους πρόσφυγες στην Ανατολική Ουκρανία και θα πρέπει όλοι μας το διάστημα που θα γίνει η συλλογή από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο, τα μέλη του Κοινοβουλίου και το προσωπικό να δείξουν δωρεία για να βοηθήσουν αυτού τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Thank you ευχαριστούμε κύριε Δίνω το λόγο στην κυρία Άννα Κορπιτσάκο που είναι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για τις παρεμβάσεις τους. Όπως ήδη υπόθηκε, η συνάντηση ανθρωπιστικού διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας οργανώθηκε την ίδια εβδομάδα με την επίσκεψή σας. Είχαμε και την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε ένα μικρό μέρος του προγραμματός σας με συμμετοχή και κάποιων από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και θεωρώ πράγματι ότι όπως και εσείς σωστά είπατε κύριε Χάουιτ, ήταν ενισχυτική η ταυτόχρονη παρουσία μας για το σκοπό μας και για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ούτως ή άλλως είχαμε την ευκαιρία να σας απενημερώσουμε για το θέμα των διαλόγων για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα σε άλλες ευκαιρίες, αλλά να πω λίγα λόγια για τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και εδώ. Για τους εσωτερικούς εκτοπισμένους και την κρίση στα ανατολικά. Μια κεχηρία στην Ανατολική Ουκρανία γίνεται σε σεβαστή περίπου από την 1η Σεπτεμβρίου και αυτό είναι θετικό για όλους όσοι κατοικούν εκεί κοντά στη γραμμή επαφής. Ωστόσο η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει τεταμένη. Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από την σύγκρουση αυτή. Όπως υπόθηκε 1,2-1,5 εκατομμύρια είναι εσωτερικώς εκτοπισμένοι στη χώρα και ο αριθμός διπλασιάστηκε από το Γενάρη. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη ευθύνη που έχει αναλάβει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Υπήρχε στο διάλογο ένα σημείο συζήτηση ακριβώ για του εσωτερικού εκτοπισμένου, Όπως το συζητήσατε και εσείς, μιλήσαμε για τους σχετικού νόμους και την εφαρμογή τους τις διαδικασίες για την αναθεώρηση των νόμων αυτών για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκε των εσωτερικών εκτοπισμένων στι χώρε. Επίσης θέσαμε θέμα για κρατική βοήθεια προς αυτούς τους ιστορικούς εκτοπισμένους, την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες, συντάξεις, επιδόματα, ε, απασχόληση και την δυνατότητα να επιβιώσουν, αλλά και να συμμετάσχουν στις επερχόμενες εκλογές. Υπάρχουν επίσης ε, ξεχωριστές ομάδες εντός της κοινότητας των εσωτερικών εκτοπισμένων, οι άνθρωποι με αναπηρίες, τα μέλη της κοινότητας των Ρωμά και το να ε, έρθουμε σε επαφή και με αυτές τις ειδικές ομάδες ε, απαιτεί εκτεκτές προσπάθειες. Κάτι που γίνεται ένα πρόβλημα και με την εξάπλωση της πολυμελίτιδας στην Ουκρανία. Από τις αρχές του μήνα συνεχίζουμε να επιμένουμε για την κύρωση, τη σημασία της κύρωσης της ε, σύμβασης για τους της Ρώμης μεταξύ και είναι σημαντικό αυτό και για την συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για το διάλογο για τα ανθρωπινιστικά δικαιώματα μας συνδράμει η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων που πρέπει να αναγνωρίσει την ε, δικαιοδοσία του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου και το οποίο σκοπό έχει εξετάσει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθησαν στην επικράτη της Ουκρανίας από τον περσινό Φεβρουάριο του 2014. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, το ίδιο και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το θέμα αυτό και το γεγονός ότι θέλουμε η Επιτροπή της Βενετίας να παρακολουθήσει και να δει την εφαρμογή των συστάσεων αυτών είναι ήδη ένα βήμα για την λογοδοσία και την αντιμετώπιση της κακομεταχείρισης και για τα θέματα των ερευνών ε, της πλατείας Μαϊντάν, για τα γεγονότα της πλατείας Μαϊντάν, για τα παράνομα κέντρα κράτησης που, ε, για τα οποία υπάρχουν καταγγελίες στον διάλογο για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Στις τοπικές εκλογές, και αυτό έχει υποθεί και από άλλε πλευρές και από την ε, Αντιπρόεδρο Μογκερίνη, Πρέπει να γίνουν λοιπόν τοπικές εκλογές στην Ουκρανία, σε όλα τα μέρη της χώρας, βάσει του Ουκρανικού νόμου και των διεθνών προτύπων. ως προς την ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να γίνουν περισσότερα Βλέπουμε πρόβλημα πρόσβαση να υπάρχει κυρίω στι περιοχέ που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει ήδη κάποια βήματα για να Διευκολύνουν τα θέματα ανθρωπιστική πρόσβαση. Η ελευθερία όμω κυκλοφορίας επίση συζητήθηκε στο διάλογο και είδαμε ότι εδώ πρέπει και εμεί και εσεί να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό πολύ προσεκτικά. Τέλο. να σημειώσω ότι ο Σαρτσένκο είναι στη Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει για να παρακολουθήσει τις συζητήσεις. Πρόεδρος. Θα ήθελα κάποιος να κάνει μια ερώτηση προς τους ε, ομιλητές για, τα, για την Ουκρανία. Όχι. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε τότε στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση για την προετοιμασία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής Κανονικά δεν έπρεπε να προεδρεύω εγώ γιατί συμπίπτω με την εισηγήτρια αυτής της έκθεσης. Δεν νομίζω τώρα ότι αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Περί πρόκειται, πρόκειται για μια αναδιαμόρφωση του ανθρωπιστικού συστήματος ε, στο ΟΗΕ που ουσιαστικά έχει εδρεωθεί πριν από 25 χρόνια και που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όμως τελείως διαφορετικές προκλήσεις. Είναι μια έκθεση για την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης και εμείς απλώς γνωμοδοτούμε ως Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο εισηγητής ο κ. Ενρίκε Γκερέρο Σαλόμ. Η ιδέα λοιπόν της διάσκεψης κορυφής για τα ανθρωπιστικά θέματα που είναι μια ιδέα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που είχε ανακοινωθεί το 2012 έχει σαν στόχο να υπάρξει πραγματικά μια παγκόσμια διάσκεψη κορυφής που θα γίνει από τις 12 ε, με 13 Μαΐου του 2016 στην Κωνσταντινούπολη και όπως σας λέω ο στόχος είναι να επικαιροποιηθεί το παγκόσμιο ανθρωπιστικό σύστημα για να μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα στις πολύ πιο πολύπλοκες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε σχέση με αυτό το οποίο ίσχυε και προβλεπόταν πριν από 25 χρόνια σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή οι ανθρωπιστικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο φτάνουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά δεν πρόκειται φυσικά για ένα οικονομικό και μόνο πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε μέσα σε αυτό το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα να κάνουμε σαφή την ανάγκη να αυξηθεί η προστασία των, των πληθυσμών και ιδίω των πιο ευαίσθητων ομάδων, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ασθενείς και συγχρόνως να δώσουμε τη δυνατότητα στους πληθυσμούς οι οποίοι έχουν πληγεί από μεγάλες ανθρωπιστικές καταστροφές ώστε να βγουν με τις δικές τους δυνάμεις από αυτή την κρίση. Είναι λοιπόν πράγματι επίκαιρη η διενέργεια αυτής της συνδιάσκεψης τη στιγμή που έχει εκραγεί ουσιαστικά η κρίση των ε, προσφύγων στις ε, χώρες της Ευρώπης. Η κρίση αυτή των προσφύγων είναι μια κρίση που υπέβοσκε σε πάρα πολλές χώρες της γειτονιά μας και σε χώρες που είναι ακόμα πιο μακριά από τα σύνορά μας, αλλά τώρα πια έχει φτάσει στα σύνορα της Ευρώπης και αυτό αύξησε την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων. Γι' αυτό εμείς ως Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε σε αυτή την έκθεση είναι να τονίσουμε ότι αυτή η αναδιαμόρφωση του διεθνούς ανθρωπιστικού συστήματος θα πρέπει να γίνει εστιάζοντας στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι απειλέ που ελοχεύουν για αυτή την προστασία και φυσικά να προστατεύσουμε και να δώσουμε τις απαραίτητες ικανότητες στα άτομα αυτά τα οποία χρειάζονται τη βοήθεια και την προστασία μας. Όπως σας είπα, η βασική έκθεση είναι από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Προθεσμία τροπολογιών τρέχει μέχρι τις 27 ε, Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και φυσικά είμαι έτοιμη να ακούσω τις απόψεις σας πάντα λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας όχι στο γενικότερο θέμα, αλλά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο μεγαλύτερο ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην δημιουργία της νέας, του νέου θεματολογίου για τα ανθρωπιστικά θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Προηγείται η ανθρωπιστική δράση οποιασδήποτε πολιτικής δράσης και φυσικά μέσα στο ανθρωπιστικό αυτό πλαίσιο μπορούμε να ενισχύσουμε την προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, δεν πριτανεύει πάντα ο σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων στην αντιμετώπιση των ε, προσφυγικών ρευμάτων ακόμα και μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα δεν υπάρχει μεγάλο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούμε να δώσουμε διδάγματα και μαθήματα στον υπόλοιπο κόσμο για το πώς να προστατεύονται οι άνθρωποι και τα ανθρωπιστικά θέματα, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα άκυρο αν τα μέσα ενημέρωσής μας δείχνουν ότι η ίδια η Ευρώπη δεν έχει κατανοήσει τι σημαίνει να προσπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι λοιπόν το κεντρικό θέμα της έκθεσης. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Ποιος έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Κόβατσεφ. Ο οποίος είναι σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ και για το σχέδιο έκθεση για την ε, ε, Επιτροπή Ανάπτυξης. Όντως, ε, είναι νέες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας και άρα χρειαζόμαστε και νέες προσεγγίσεις. Καλωσορίζουμε την Σύνοδο, θα τον πρωτοβουλία Γενικού Γραμματέα ε, του ΟΗΕ. Φυσικά πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και να καταβάλουμε ε, ισχυρότερες προσπάθειες ε, και στον τομέα της παιδείας. Σε επίπεδο διεθνούς κοινότητα επίσης θα πρέπει να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η εμπορία ανθρώπων, η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ε, ε, ομάδων, η στρατολόγηση ανθρώπων σε αυτές τις, ε, σε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις, στρατολόγηση αλλοδαπών μαχητών και το καθεξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να πάψει η χρηματοδότηση οργανώσεων όπως το Ισλαμικό κράτος. Και φυσικά η πολιτική η ισότητα των δύο φύλων δεν είναι κεντρικό μεν ζήτημα, απαραίτητο δε για να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις διαστάσεις του ζητήματος. Σε παιδεία, όπως σας είπα, ένα με σημαντική προτεραιότητα. Διαθεσκευτικός διάλογος. Εμείς το ΕΛΚΑ θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε και πάλι και θα σας υποστηρίξουμε. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Μπεσέρα, που είναι η συγγήτρια εισηγήτρια εκ μέρου του Σάλντε και για να αποτιμήσουμε μαζί την έκθεση που μόλις μας παρουσιάσατε. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την εισηγήτρια την κυρία Βαλεντιάνου για αυτή την τόσο διεξοδική έκθεση που καλύπτει τόσες πολλές ε, καθοριστικές πτυχές της ανθρωπιστικής μας πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το κείμενο υπάρχουν οι τροπολογίες μου με στόχο να διασυνδέσουμε συγκεκριμένε δράσεις της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις σχετικές χάρτες του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για μια δικαιολόγητη δήλωση ή αφηρημένη, αλλά στόχο οι καταλληλές προϋποθέσεις και όροι να προσπαθούν στους πρόσφυγες για να έχουν μια κανονική ζωή Άρα η σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, σχετικές υπηρεσίες και η δέσμευσή μας προς μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε καιρούς ανθρωπιστικής κρίσης είναι κάτι που πρέπει να γίνει σεβαστό ταυτόχρονα. Οι δεσμεύσεις μας με την παροχή υγειονομικών ε, υπηρεσιών και πόσιμου νερού για να αποφευθεί επιδημία είναι πολύ σημαντικά ακρογωνίως λήθος για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα στη ζωή και την αξιοπρέπεια. Λόγω χάρη πρόσβαση σε φάρμακα και υγειονομικές υπηρεσίες είναι ένα πρόβλημα που συχνά αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Η παροχή αυτής της υπηρεσίας δεν έχει να κάνει μόνο με το να δοθεί βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μαζί με όλες τις άλλες πτυχές της ανθρωπιστικής μας δράσης έχουν να κάνουν με κάτι παραπάνω από την ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ότι στόχος της ανθρωπιστικής πολιτικής είναι να δίδεται η ευθύνη για την κατάστασή τους στα ίδια τα ανθρώπινα όντα για να ξεπερνάνε τις δυσκολίε. Αυτή η εξουσία έχει να κάνει με την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Έχει να κάνει με την δυνατότητα, την ευκαιρία, την δραστήρια στάση ενός ανθρώπου που μπορεί να προχωρήσει, να πετύχει και να εκπληρώσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Όταν αυτά μπορούν να λειτουργήσουν υπάρχει η περίπτωση να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αρκεί. Αυτός ο δρόμος ε, είναι ε, μόνο η αρχή και προς αυτήν την κατεύθυνση δεσμεύομαι και ο ίδια. Στηρίζω την ε, τοποθέτηση αυτή. Ευχαριστούμε κύριο Ντεμεσμέκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Βαλεντιάνο. Από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το έργο που έχετε φέρει σε πέρας για την έκθεση αυτή. βλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας. Ο σκιώδης μας δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε 60 εκατομμύρια προσφύγων σε όλο τον κόσμο Είχαμε προηγουμένως τη συζήτηση για την Ουκρανία που είδαμε ότι πρόκειται για 5 εκατομμύρια ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική δομή, βοήθεια 1,5 εκατομμύριο ατόμων εσωτερικά εκτοπισμένων. Είναι τεράστιες λοιπόν προκλήσεις που έχει ενώπιον της η διεθνής ε, ανθρωπιστική κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά μόνη δεν μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε συγχρόνως η διάσκεψη αυτή να γίνει μοναχά μια λέσχη συζητήσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα προκύψουν και κάποια αποτελέσματα από τη διάσκεψη Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Το, το αποτέλεσμα θα εξαρτάται από το αν θα υπάρξουν νέοι συνομιλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διάσκεψη. Γιατί πιστεύω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗ ήθελε να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι από τις επιτόπιες οργανώσεις. Αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μονάχα μία διάσκεψη η οποία θα έχει καθαρά διακυβερνητικό χαρακτήρα. Θα ήταν χρήσιμο να γίνει κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια πραγματική αντιμετώπιση της κρίσης. Και ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ τη Ανθρωπιστική Βοήθεια Κομισιόν δηλαδή. Η πρώτη χωρί μικρόφωνο. Θα μας πει η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ που εκπροσωπείται εδώ. Ο κύριος Βόλφκαν Στρέιτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας να σα ευχαριστήσω για την διεξοδική σα τοποθέτηση και όλου του ε, βουλευτέ για τη συνεισφορά του στη συζήτηση. Είμαι βέβαιο ότι πολλά από τα θέματα που θίγετε στην κομμοδότησή σα θα συνεχίσουν να συζητώνται όλη τη χρονιά αυτή στο Κοινοβούλιο και μετά τις προπαρασκευαστικέ δραστηριότητε ε, για το κείμενο τη διάσκεψης. Να σα θυμίσω απλώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε μια ανακοίνωση για αυτή την παγκόσμια συνεδοκορυφή Υπάρχει και σχετικό φυλάδιο για το ζήτημα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν προσπαθήσαμε να καθορίσουμε τη θέση μα εν ώψη της Συνόδου και να κάνουμε συγκεκριμένε συστάσεις με τομείς προτεραιότητας. Νομίζω για το σκοπό του έργου της δικής σας Επιτροπής θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ανακοίνωση επικεντρώνεται στην ε, ε, ανθρωπιστική δράση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος από τη δική σας τη Σκοπιά η πιο σημαντική τομής ήταν ο τομέας 1 για τις ανθρωπιστικές αξίες, τις ουδετερότητας αμεροληψία, ανεξαρτησία και ανθρωπιάς, καθώς και ο τομέας 3 όπου θα θέλαμε η διάσκεψη την προστασία να την βάλει στον πυρήνα των του συστήματος ανθρωπιστικών ε, αποκρίσεων. Εκεί η συζήτηση περί ανθρωπιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικά ε, συνενώνονται και καταλήγουμε στο κλίμα που θα πρέπει να επικρατήσει στη διάσκεψη. Ακούσαμε προσεκτικά τη συζήτησή σας για τη Γάζα και την ε, Ουκρανία και φαίνεται ότι το έργο της Επιτροπής σας ε, πραγματικά παρακολουθεί την εξέλιξη των ανθρωπιστικών ζητημάτων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά και χρήσιμα στοιχεία. Παρατηρήσεις για την εκπαίδευση, όπου σκοπεύουμε να εντείνουμε τη χρηματοδότησή μας για αντιμετώπιση κατεπίγουσων καταστάσεων. Οι προτεραιότητες και αντιμετώπιση της βασισμένης στο φύλλο και δύο παρατηρήσεις πρωτού κλείσω. Ε, η διακυβερνητική προσέγγιση που ζητάτε και σε σχέση με το κείμενο για τη διάσκεψη να θυμίσω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ έχει καθορίσει μια ανοιχτή πορεία που συμπεριλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, τις κυβερνητικές οργανώσεις και κατοικούς φορείς δεν πρόκειται για κυβερνητική διάσκεψη που θα αποφασίσει απλώς η συνέχεια της Συνόδου Κορυφής δεν θα πάρει μάλλον επίσημη μορφή μέσω του μηχανισμού, των μηχανισμών των Ηνωμένων και μετά θα εκφραστεί και σε κυβερνητικές αποφάσεις. Διακυβερνητικές μάλλον αποφάσεις. Όπω τι αρχέ που θα είναι η βάση για τι ανθρωπιστικέ ε, δράσει και η επόμενη διάσταση που είναι η προσέγγιση βασισμένη σε ανάγκες αυτό προσπαθούμε να ακολουθήσουμε γιατί είμαστε φορεί που εξασφαλίζουν προστασία και εγγυώνται το ανθρωπιστικό δίκαιο παγκοσμίω πιστεύω, αυτό είναι σαφέ στα προγράμματά μας, αλλά θα θέλαμε να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί για το πώς μπορούμε να μετρώμε τις ανθρωπιστικέ δράσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, συνέχεια, ε, που συνήθως είναι στα χέρια κυβερνητικών φορέων ή αναπτυξιακών έστω φορέων. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Ξέρετε ποια είναι η προθεσμία για τροπολογίας. 24 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω ότι υπάρχουν εδώ παρόντες εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ακόμα και αν λείπουν οι συγητές, ξέρουμε ότι μέχρι τότε είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συζήτηση που μπορεί να βελτιώσει την γνωμοδότηση αυτή. Και τώρα εκεί. Κίνη η συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρίου. Παρακαλώ να μείνουν στην αίθουσα μόνο οι αντιπρόεδροι και οι συντονιστές και το κοινό θα πρέπει να αποχωρήσει.